Dear members and... Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί καλεσμένοι, καλησπέρα σας. Head of Secretariat is telling me that there is... Ο γραμματέας μου επισήμανε ότι είναι στη διάθεση του προσωρινού προέδρου και το σφυράκι. Ε, ελπίζω να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω όμως. Ε, ήδη έχουμε μια τετράλεπτη καθυστέρηση. Γι' αυτό παρακαλώ καθίστε το συντομότερο για να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ θερμότατα και ειλικρινέστατα και το, τα παλιότερα μέλη που έχουν επανακλεγεί, αλλά και τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της ΙΝΤΑ. Καλώς ήρθατε λοιπόν θερμά. Πρόκειται για την, την συνεδρία συγκρότηση σώμα αυτής της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΙΝΤΑ και εγώ ως απερχόμενος ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ ορίστηκα ως προσωρινός πρόεδρος της ε, Επιτροπής. Και όντως θα είναι πολύ προσωρινή η προεδρία μου, γιατί το μόνο μου καθήκον είναι να προεδρεύσω κατά τη διάρκεια της εκλογής του νέου Προέδρου. Και αμέσως μετά, μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, θα δώσω τη σκητάλη στον νέο Πρόεδρο για να προεδρεύσει. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασης και να σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Καταρχάς, ο σκοπός της συνεδρίασης αυτής είναι ένας και μόνο. Να συγκροτήσουμε σε σώμα την Επιτροπή και να, ε, εγκρίνουμε με βάση το άρθρο 213 της, του εσωτερικού κανονισμού τον Πρόεδρο και τους α, Αντιπρόεδρους της Να στήσουμε δηλαδή το Προεδρείο. Πρώτα φυσικά θα εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, την πρόεδρο και μετά τους αντιπρόεδρους. Και πριν να προχωρήσουμε θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας γιατί πολύ πιθανό να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε. Αν την ξεχάσατε στείλτε κατεπηγόντως κάποιον ε, βοηθό να σας τη φέρει. Έχω και ένα κατάλογο μαζί μου, γιατί δεν είναι μόνο... Δεν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, οπότε θα τους αναπληρώσουν τα αναπληρωματικά μέλη. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αναπληρώτρια. Αναπληρώ... Αναπληρώνεται από τον κύριο Γιώτας Μάσλης. Δανιέλ Κασπάρη, τον αντικαθιστά, τον αντικαθιστά η Άννη Πύρικ και η Διουριάνικε αντικαθίσταται από, τη... από τον Λόραν Γιοντβίντσε. Από το ΕΛΚ ήταν αυτή και από το ECR η Βαρόνη Μόμπαρικ αντικαθιστά τον Κυριάκο Βελόπουλο που είναι τακτικό μέλος της ΣΥΝΤΑ. Αυτές ήταν ε, οι ανακοινώσεις για κάποιες αντικαταστάσεις τακτικών από Α Έχουμε και μια άλλη ακόμη αντικατάσταση. Ο κύριο Σούστερ από του και Δημοκράτε αντικαθιστά τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι επίση τακτικό μέλος τη Επιτροπής Ίντα. Έχουμε πέντε δηλαδή αναπληρωτές που αντικαθιστούν τακτικά μέλη και αν κάποια πολιτική ομάδα θέλει να προβεί σε καμία ανακοίνωση για άλλες αντικαταστάσεις, δεν βλέπω, οπότε περνάμε στο πρώτο κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Καταρχήν να επιβεβαιώσω ότι ε, υπάρχει απαρτία, άρα θα είναι έγκυρη η ψηφοφορία. Έχουμε πάνω από 11 μέλη παρόντα από την Επιτροπή Ίντα. Έχουμε τον κατάλογο, οπότε απαρτία υπάρχει. Και τώρα, βάσει του εσωτερικού κανονισμού, θα ήθελα να ε, ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την θέση του Προέδρου της ΣΥΝΤΑ. Κυρία Βαμπρέντα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα του Μπέντ Λάγκε για την Προεδρία της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την υποψηφιότητα του Μπέντ Λάγκε για τη θέση του Προέδρου. Άλλες πολιτικές ομάδες έχουν να προτείνουν υποψηφίους για, το, για την Προεδρία της ΣΥΝΤΑ. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ο, ο κύριος Μπέρντ Λάγκε, ο υποψήφιος, δέχεται τη, την υποψηφιότητά του. Βεβαίως ε, και με τιμά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνένεσή σας. θέλετε κάποια ιδιαίτερη μορφή ψηφοφορίας. Δεν έχει υποβληθεί γραπτό αίτημα για ειδική ψηφοφορία, απλώς το τσεκάρω με τα μέλη της Επιτροπής δεν έχει υποβληθεί έτοιμα για κάποια ειδική μορφή ψηφοφορίας, οπότε ως ήθιστε θα εκλέξουμε διαβοή στον υποψήφιο, τον κύριο Μπέρντ Λάγκε. Οπότε ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Επιτροπής Σύντα καλείται να έρθει και να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής. So, Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εκλογή, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι εκ νέου πρόεδρος της ε, πολύ σημαντικής ε, εξαιρετικής αυτής επιτροπής, μια σημαντικής επιτροπής για το Κοινοβούλιο και είμαι πεπισμένος πως θα συνεχίσουμε το έργο μας σίγουρα θα δίστανται απόσμα σε κάποια ζητήματα. Όπως όμως κατά το παρελθόν καταφέραμε να συνεργαστούμε πολύ καλά, το ίδιο θα πράξω και αυτή τη θητεία. Ε, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την εμπορική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο μια καλύτερη και πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Σας ευχαριστώ θερμά εκ νέου λοιπόν και θέλω θερμά να καλωσορίσω ιδίως ε, τα νέα μέλη αυτής της Επιτροπής. 30 από τα 41 μέλη της Επιτροπής μας είναι νέοι συνάδελφοι. Οι σαρπαστικοί ενδιαφέροντες και νέες φρέσκες ιδέες και όλα αυτά τα θεωρώ ιδιαίτερα θετικά. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου καταρχάς. Ο κύριος Βίνκλερ ανέφερε τον κατάλογο των ε, αντικαταστατών από των συναδέλφων. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ακούσω ψηφιότητε για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξανόματο ομάδος ομάδα του ECR θα ήθελα να προτείνω ω υποψήφιο τον κύριο Γιάνν Ζάχραντιλ. Νομίζω είναι γνωστός από τους ευρωβουλευτές. Ε, έχει μακρά εμπειρία και είναι ανοιχτός ε, για έναν επικοδομητικό διάλογο και θέλει και ένα διεθνές εμπόριο βάση κανόνων. Τέλεια, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Από ό,τι βλέπω όχι. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κ. Ζαχράντιλ να μας πει κατά πόσον επιβεβαιώνει την υποψηφιότητά του κύριε Σαχράτλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη τιμή αποδέχομαι και θα συνεχίσω να υπηρετώ την Επιτροπή αυτή ως αντιπρόεδρος εφόσον εκλεγώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, τέλεια. Επομένως έχουμε έναν μόνο υποψήφιο ο οποίο συμφωνεί με, την, με τον ορισμό και προτείνω να τον εκλέξουμε διαβοής. Thanks a lot, Mr. Sadiel. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαχράντιλ. Καλή συνεργασία. Ελάτε εδώ, ελάτε σε μένα κύριε Ζαχράντιλ. Thank you, Mr. Chairman. Hi, good So, next item is Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου και παρακαλώ τώρα να ακούσουμε τις υποψηφιότητες για την θέση αυτή. Mr. Chair, may I interest you in... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υποβάλω στην υποψηφιότητα τον κύριο Μαξιμίλιαν Κράχ από το ΙΔ, e που σπούδασε νομική στη Γερμανία και έχει πάρει και ε, διδακτορικό για ε, ένα ζήτημα έχει εργαστεί και σε ένα MBA στο Κολούμπια και στο LSE. Έχει εργαστεί και στο πλευρό του Στίγκλιτς ε, και είναι εταιρικό δικηγόρο, υπήρξε μέλο ΔΣ σε χώρε όπω η Λετωνία, η Αυστρία και στη Γερμανία ε, εξελέγει πρόσφατα Ευρωβουλευτής. Και νομίζω ότι λόγω του ακαδημαϊκού επαγγελματικού υποβάθρου του είναι ο κατάλληλο για αυτή τη θέση. Θα προαγάγει ελεύθερη ροδιάλογο, ε, συνεργασία. Θέλω να σας ε, πενθυμίσω και τον κανόνα 213 που λέει ότι πρέπει να υπάρχει πολυμορφία ε, όπως υπάρχει στο Κοινοβούλιο και αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση των Προεδρίων. Νομίζω ότι όλα αυτά θα είναι προς όφελός μας, αν εκλέξουμε τον κύριο Κρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Βίνκα να συνεχίσει στη θέση του Αντιπρόεδρου, τον ξέρετε. Τον έχετε συναντήσει. Και ήταν εκείνο που κήρυξε και την έναρξη. Νομίζω ότι είναι πολύ ικανό και με χαρά θα σα ε, στηρίξει στη δουλειά σα ε, ω αντιπρόεδρο. Κύριο Λάγκεν, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Όχι. Παρακαλώ λοιπόν τους δύο υποψηφίους μας να έρθουν. Κύριε Καν, συμφωνείτε, δέχεστε καταρχάς. Μάλιστα, κύριε Βίνκλερ. Πρόεδρε και συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την ομάδα μου από το ΕΛΚ για την ε, προβολή της υποψηφιότητά μου. Καλώς, έχουμε δύο υποψηφίου λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. So, my secretariat said I have to... Η γραμματεία μου λέει ότι πρέπει να σας εξηγήσω επακριβώς τη διαδικασία ψηφοφοριών. Έχετε λοιπόν μία ψήφο έκαστος και εκάστη. 10 από το ΕΛΚΑ, 9 από τους ΕΛΣΤΕΣ, 6 από το ΑΛΔΕ, 3 από την 1, μία εγγεγραμμένη 3, και όποιος έχει την απόλυτη πλειοψηφία, όποιος κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, Συνεχίζω με τους Γκουε που έχουν δύο ψήφους, πράσινοι έχουν τέσσερις, το Renew Europe έχει έξι ψήφους. Και... Όποιο κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται, αλλά η απόλυτη πλειοψηφία διαφέρει από αυτό που έχουμε στον Αμέλεια, γιατί δεν μετράνε οι αποχές για τον υπολογισμό της απόλυτης πλειοψηφίας. Everybody should have Έχετε όλη την κάρτα σας, την ηλεκτρονική. Τα ονόματα είναι γνωστά. Για να βάλουμε και ένα χρώμα λοιπόν στον κάθε υποψήφιο. Πράσινο, άσπρο, κόκκινο, τι θέλετε, ο κύριος Βίνκλερ. Πράσινο λέει. Να πούμε τότε κόκκινο για τον κύριο Καν. Κάνουμε δοκιμαστική πρώτα ψηφοφορία και παρακαλώ θα είναι αυτό ευκαιρία να δοκιμαστεί η κάρτα στο μηχάνημα. Αρχίζουμε. Έχουμε έναν υπεράριθμο strange. But only 38 have voted, so uh, One too many. it doesn't matter. So we have 42 members with a card. 42 έχουν βάλει κάρτα στο σύστημα, αλλά 39 μόνο επιτρέπεται να ψηφίσουν. Παρακαλώ, όποιος και όποια, ας επαληθεύσετε. Και μάλιστα τώρα γίνανε 43 οι κάρτες. Εδώ δυστυχώς το μηχάνημα που έχω δεν μου επιτρέπει να δω από ποια ομάδα είναι η κάρτα, οι υπεραριθμές κάρτες. Επαληθεύστε παρακαλώ. Οι πολιτικές ομάδες παρακαλώ να επαληθεύσουν. 10 το ΕΛΚ. 8 οι σοσιαλιστές δημοκρατές. 8. 6 το Renew Europe. 4 οι πράσινοι. 5 το ID. 3 το ECR. GUNGL 2. Μία εγγεγραμμένη τρεις. Μία, δύο, τρεις. Καλά, τότε δεν ψηφίζω εγώ. Και γύρω ένα 41. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Επαληθεύουμε πρώτα. Η εποχή είναι το άσπρο στη μέση. Πρόεδρε, επαναλαμβάνετε παρακαλώ τα χρώματα. Ο κύριος Βίγκλερ έχει το πράσινο. Ο κύριος Κά έχει το κόκκινο. Το λευκό είναι η εποχή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Κύριε Γκριν. Κύριε Βίνκλερ. Εκλεγήκατε, κύριε Πράσινε. Το δέχεστε, μάλιστα και ευχαριστώ. Then Επόμενο σημείο, η εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Ποιοι είναι οι υποψήφοι για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη θέση της τρίτης αντιπρόεδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Η κυρία Σιμακοπούλου δυστυχώς ακολύεται και απουσιάζει. Θα διαβάσω όμως μία δήλωσή της για την υποψηφιότητά της. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Καταρχήν θα ήθελα να σα ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για την απουσία μου. Αλλά ε, οι ελληνικέ εκλογέ που προηγήθηκαν με εμπόδισαν να έρθω εδώ κατά την εκλογή των αντιπροέδρων και με μεγάλη τιμή θα δεχτώ την ψήφα εμπιστοσύνη που θα μου δώσετε, αν θα μου τη δώσετε και θα ε, εργαστώ με αποφασιστικότητα και αφοσίωση για να προτάξω τις προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Διεθνές Εμπόριο και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας. Μάλιστα, μας έγραψε και μια δήλωση ότι συμφωνεί με τη διαδικασία. Ε, θα ήθελα και πάλι να προτείνω την υποψηφιότητα του κύριου Μαξίμιλιαν Κρά για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως ε, για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν. Όχι κύριε Κά, δέχεστε την υποψηφιότητα, μάλιστα. Οπότε θα ισχύσει η ίδια διαδικασία. Ας κρατήσουμε τα ίδια χρώματα, δηλαδή το πράσινο χρώμα για την υποψήφια του ΕΛΚ, την κυρία Σημακοπούλου, και το κόκκινο χρώμα για τον κύριο Κα, τον υποψήφιο του ID, και λευκό χρώμα ή αποχές. Άρχεται οι ψηφοφορία. And the Τέλος Η υποψήφια του ΕΛΚ εκλέγεται. Στείλτε στις τα συγχαρητήρια παρακαλώ. Και περνάμε στην εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Και ρωτώ, υπάρχουν υποψήφοι για αυτή τη θέση. Μάλιστα. Με χαρά θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα της κυρίας Μαρή Πιέρ Βοντρέν. Η Μαρή Πιέρ είναι Γαλλίδα, 63 ε, ετών. Είχε μάστερ στο δίκαιο του ΠΟΕ. Γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα και το διεθνές εμπόριο και διατέλεσε και ε, διευθύντρια για τέσσερα χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οίκο τη ΡΕΝ και μάλιστα είχε στενέ επαφέ και συχνέ επαφέ με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για θέματα εμπορίου, ιδιαίτερα ε, εμπορικές σχέσεις με τι Ηνωμένες Πολιτείες και συμφωνία ΣΕΤΑ με το Καναδά. Εκ μέρου της ομάδας ε, Renew θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα της ε, Μαριπιέχα Ντατρέν. Άλλοι υποψήφοι υπάρχουν, παρακαλώ, για τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ. Όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε ερωτώ την μία και μοναδική υποψήφια αν συμφωνεί. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, με τιμά ιδιαίτερο αυτή η πρόταση και τη δέχομαι ευχαρίστω. Λαμπρά. Έχουμε μόνο μία υποψήφια, οπότε μπορούμε να την εκλέξουμε διαβοής. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να έχουμε πολύ καλές ε, σχέσεις και συνεργασία στην κοινοβουλευτική μας θητεία. Είμαι τώρα στο σημείο 6 της της διάταξης. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Πρώτο θέμα, η πρόταση για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων μας για το 2019 έχετε λάβει στους φακέλους σας την πρόταση για τις ε, ημερομηνίες συνεδρίασης. Έχω και μία επιπλέον παρατήρηση. Πολλές ομάδες ζήτησαν να προσθέσουμε μία συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου. Θα εφαρμόσουμε τη γραπτή διαδικασία με τους συντονιστές ώστε θα γνωρίζετε μέχρι την Τρίτη αν θα οργανωθεί και επιπλέον μία επιπλέον συνεδρίαση. Ο βασικός στόχος της συνεδρίας αυτής, Αργίνη, θα είναι η συνεδρίαση με τον, επίτροπο, τον αρμόδιο επίτροπο για το Μερκοσούρ. Οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων με την πιθανότητα για μια επιπλέον συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου. Υπάρχουν αντιρρήσεις στο σχέδιο προγράμματος των συνεδριάσεων. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σε συγχαρώ, Μπέρντ, για την εκλογή σου και φυσικά και τους αντιπρόεδρους το ίδιο. Είχαμε ήδη ευκαιρία στο παρελθόν να συνεργαστούμε στενά και προσβλέπω σε πολύ επικοινωνητικό διάλογο και καρποφόρα συνεργασία στο μέλλον. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την εργαστή συνεργασία. Καθήκον σου είναι να εκπροσωπείς την πολυμορφία της Επιτροπής μας και προς τα έξω. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι για την εντολή που ανέλαβες. Για το πρόγραμμά μας, το χρονοδιάγραμμα, βλέπω ότι έχουμε συνεδριάσεις που ξεκινά στις 2.30. Είναι απολύτως απαραίτητο. Προτιμούμε να ξεκινούν στις 3 το απόγευμα οι συνεδριάσεις, όχι στις 2.30 και αυτό το αλλάξαμε και πριν τι εκλογέ. Αυτό το κάναμε πριν τι εκλογέ, γιατί είχαμε πολλές, πολλά θέματα. Οπότε προτείνω αυτή την αλλαγή. Για το Μερκοσούρ χαίρομαι που προτείνατε μια επιπλέον συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να υποφασίσουμε και σήμερα, αφού είναι παρόντε οι συντονιστέ, να δούμε αν συμφωνούν. Να προσθέσουμε μια επιπλέον συνεδρίαση στι 23 Ιουλίου για το Μερκοσούρ. Και αρχικά είχε προβλεφθεί η συνεδρίαση αυτή, δεν είναι καν συμπληρωματική. Οπότε α αφήσουμε τη συνεδρία τη 23η που υπήρχε αρχικά. Ελπίζω να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι συντονιστέ και να ε, ζητήσουμε εγκαίρω ε, από την Επίτροπο να έρθει, γιατί έχει περφορτωμένο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι συντονιστέ τη γνώμη έχουν η κυρία Μπρέμπτ. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κύριε Λάγκη για την εκλογή σα και ε, φυσικά συγχαρητήρια και στου άλλου αντιπροέδρου. Είστε πολύ ικανό. Εγώ είμαι καινούργια βέβαια στην Επιτροπή Ιντα. Πάντω έμαθα ότι η προηγούμενη πενταετία ήταν πολύ επιτυχής για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Προσβλέπω λοιπόν σε στενή συνεργασία και ανοιχτό συντονισμό, όπως γίνεται σε αυτή την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, συμφωνώ με την πρότασή σα να εφαρμοστεί η γραπτή διαδικασία μεταξύ των συντονιστών, γιατί έχουμε πολλά νέα μέλη στην Επιτροπή μα, όπω είπε και ο Πρόεδρο προηγουμένω, ειδικά στην ομάδα μου. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για διαβουλεύσεις και επί του προγράμματος και επί του περιεχομένου. Οπότε προτιμώ τη γραπτή διαδικασία που προτείνατε αρχικά. Μάλιστα. Η φιλελεύθερη. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια φυσικά στον πρόεδρο και στους αντιπρόεδρους. Και εμείς ε, αδειμονούμε ε, να ξεκινήσουμε τις εργασίες και την συνεργασία μας. Είναι πολύ καλή να προσθεθεί η συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου, γιατί πολλοί είμαστε καινούργοι και θέλουμε να κατατοπιστούμε όσο γίνεται περισσότερο πριν τις θερινές διακοπές. Και από ό,τι ξέρω και η Επίτροπος Μάλμστρο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και θα δεχτεί ευχαρίστω την πρόσκληση στη συνεδρίαση αυτή. Ελπίζω να συμφωνήσουμε και να προσθεθεί αυτή η συνεδρίαση τη 23 η Ιουλίου. Ε, από τους πράσινους ποια είναι η συντονίστρια, η Χάιδη Χάουταλα. Ναι, Μπορούμε να δεχθούμε την ε, πρόταση σας για την ε, γραπτή διαδικασία. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζω στη μετρική μου γλώσσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και να σας συγχαρώ και τους αντιπροέδρους για την μελλοντική συνεργασία όσον αφορά το πρόγραμμα. Προτείνω να ακολουθήσουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Να έχουμε αυτή τη συζήτηση στις 23 του μηνός. Είναι σημαντικό το θέμα. Εγώ δεν σας συγχαίρω, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έγινε παρουσίαση. Δεν καλύπτεται μάλλον η... Ε, ποικιλία που απαιτείται και θα έπρεπε το ΕΛΚ να ντρέπεται για την εκπροσώπηση αυτή στο ε, Προεδρείο. Γκουε. Κύριε Λάγκα, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια σε εσά και του συναδέλφου σα. Δεν ορίστηκε ακόμα συντονιστή από την ΚΟΕ, Πάντω. αφού είμαστε μόνο δύο, δεν θα είναι δύσκολο, Σα καθησυχάζω. Καλώ ήρθατε οι νέοι συνάδελφοι αν θέλετε στις 23 Ιουλίου ε, συνεδρίαση για να ζητήσετε από την κυρία Μάλστρομ πληροφορία για τη Μερκοσούρ. Εντάξει, αλλά να μην βιαζόμαστε κιόλα, γιατί έχουμε ακόμα δύο χρόνια μπροστά μα. Δεν τελειώνει το θέμα πριν το καλοκαίρι. Και έχουμε πολλά επιχειρήματα. Είτε κάνουμε τη συνεδρία 23 Ιουλίου, είτε όχι. Η συζήτηση για τη Μερκοσούρ, αλλά και για όλα τα άλλα, γιατί έχουμε και την εκθέση για το Βιετνάμ που θα πρέπει να κυρωθεί πριν από το τέλο του 19. Θα μα βρουν παρόντες. So the coordinators are split. Um, therefore I really propose to have a really written Καλώς, επομένως, διαδικασία γραπτή, όχι, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν μέτρησα καλά, αλλά... τρία, τρεις ομάδες, Renew, ECR, EPP, έχουν ε, στηρίξει. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πλειοψηφία. Ναι, εμείς συμφωνούμε να ξεκινήσουμε στις 23 τη διαδικασία για την ε, συνθήκη Μερκοσούρ. Καλώς λέει ο πρόεδρος, τώρα ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Υπάρχει πλειοψηφία λοιπόν υπέρ της επιπλέον αυτής συνεδρίασης για τις 23 Ιουλίου αλλά ελπίζω οι ομάδες που ήταν υπέρ της συνεδρίας αυτής και είπαμε ότι δεν θα έχουμε τίποτα καινούριο, σωστά το είπε ο Μανουέλ. Ελπίζω λοιπόν οι ομάδες να μεριμνήσουν να υπάρχουν εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση. Όταν ζητούμε συνεδρίαση πρέπει να έχουμε και παρουσίες. Μετά ο κύριος Φάνης έκανε μια άλλη, συνεδρία, μια άλλη πρόταση οι συνεδριάσεις να ξεκινούν όχι στις 2.30 αλλά στις 3. Νομίζω ότι πολύ εύστοχα το προτείνει. Είχε γίνει μια αλλαγή στα τέλη της προηγούμενης ε, θητείας, γιατί είχαμε πολλή δουλειά και έπρεπε να τελειώσουν τα θέματα. Αλλά βεβαίω τώρα πια μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα καθιερωμένα και να ξεκινούμε στις 3 το απόγευμα, οπότε θα έχουμε και πιο πολύ χρόνο για το μεσημεριανό μας. Αυτά. Έχετε κάτι άλλο? Άλλες παρατηρήσεις για το σχέδιο χρονοδιαγράμματος για το δεύτερο ήμιση του 19. Εγκρίνεται λοιπόν. Δεύτερη ανακοίνωση. Υπάρχει ένα ε, πακέτο υποδοχής για όλους σας ε, που σας δείχνει, σας δίνει πληροφορίες για τον τρόπο λήψη αποφάσεων, γενικά για τις διαδικασίες εδώ στην Επιτροπή μας. Θα το βρείτε στα, ε, στις εκδρομικές αστερίδες στον τρίτο όροφο. Επίση, εξουσίες για τους συντονιστέ, άλλη απόφαση που έχουμε να λάβουμε. Ξέρετε ότι με βάση το άρθρο 214, παράγραφο 2 του ιστορικού κανονισμού, οι συντονιστέ προετοιμάζουν τις εργασίες και τις αποφάσει που καλείται να λάβει η Επιτροπή. Και σε αυτούς εκχωρείται από την Επιτροπή η σχετική εξουσία. Είναι καθιερωμένη η πρακτική στην Επιτροπή μας αυτό και έτσι θα ήθελα να εκχωρηθούν στους συντονιστές μας, με κάποιες εξαιρέσεις ασφαλώς, οι σχετικές εξουσίες, εκτός από την έγκριση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, προφορικών ερωτήσεων που θα πρέπει να ψηφίζονται εδώ στην Επιτροπή στην πλήρη τη σύνθεση. Σχόλια έχετε για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους συντονιστές. So then, um, if there are no objections to this proposal, δεν βλέπω αντιρρήσεις. Εγκρίνουμε λοιπόν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων για να ξεκινήσει η δουλειά. Πέμπτη πρωί την επόμενη εβδομάδα μπορεί να γίνουν η συνεδρία των συντονιστών στο Στρασβούργο. Επίση, δεν έχουν υπογράψει όλοι οι συνάδελφοι τον κατάλογο παρουσιών. Παρακαλώ, μην το λησμονείτε. Γιατί είναι σαφής απόδειξη της παρουσίας εδώ. the most liked item, uh, for... Και ένα τελευταίο. τριμερή σε διάταξη που έχει λησμονηθεί. Είναι τα διάφορα. Διάφορα λοιπόν. Έχετε κάτι για τα διάφορα. Και πάω στο 7, γιατί τα διάφορα ήταν το 8. Η, μερίσια, ε, η προσεχή συνεδρίαση 23 Ιουλίου πρωί, 9 η ώρα.